τα ε, όσα εγκρίθηκαν στην προηγούμενη σύνοδο ε, και θα είναι διαθέσιμα για όλους σας από το ΕΛΚ και από τους Πράσινους από την ε, Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία έχω τα εξής να σας πω σε σχέση με τις κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και θα δείτε τον κατάλογο αυτών των διορισμών στη πρακτικά αυτή της ε, συνόδου. Εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται αυτοί οι διορισμοί στις κοινοβουλευτικέ ομάδες. Και τώρα περνάμε στην ημερήσια διάταξη της Συνόδου, τις τέσσερι μέρες δηλαδή τη Συνόδου, το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης